Chers amis, bonjour. Je vous propose d'ouvrir notre. Αγαπητοί φίλοι, προτείνω να ξεκινήσουμε τις ε, δύο ώρες συζητήσεων για το θέμα των σχέσεων μεταξύ mm. Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Αρμενίας διορθώνει η Πρόεδρος. Ξέρετε, είναι και εκτιμένη ταχύτητα λόγω της ε, θέσεώς μου. Σχέσεων, λοιπόν μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Καλώς ορίζω όλους τους παρόντες και ιδίω. θα ήθελα να πω ότι έχουμε τη Ρακέλ Ντίνκ παρούσα. Μας θύμισε χτες με την ε, εγγενίαση της εκθέσεως του Ιδρύματος Χραντίνκ το οποίο μπορείτε πάντα να επισκεφθείτε, είναι στο ισόγειο του Κοινοβουλίου. πέντε ταινίες σύντομες οι οποίες έχουν γυριστεί γύρω από το θέμα της καθημερινής ζωής, τα σύνορα αυτά, τουρκο-αρμενικά σύνορα που έχουν κλείσει, παραμένουν κλειστά τα οδικά σύνορα από το 1993. Και θα είναι το αντικείμενο τη σημερινή μα συνεδρία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων και επίση θα πρέπει να σημειώσω ε, την ε, συγνώμη του Προέδρου της ε, εν λόγω Επιτροπής ο οποίος για λόγους που πιστεύω είναι κατανοητοί και που αφορούν την πατρίδα του, δηλαδή τις εκλογές στη Γερμανία, δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρόν, και της αντιπροσωπείας για τη σχέση με τον ε, Νότιο Κάφκασο, ο φίλος Μίλαν είναι δίπλα μου, καθώς και της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Τουρκία. Η συζήτηση αυτή στηρίζεται σε δύο κείμενα αναλογισμού και αναλύσεως και προτάσεις. Δύο τοποθετήσεις που ζητήσαμε σε δύο ειδικού εμπειρογνώμονες ε, γνώσεις της καταστάσεως, τον κύριο Τζέγκη Ακτάρ, ο οποίος είναι καθηγητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, και τον κύριο Ρίτσαρτ Τύραγκος ο οποίος είναι Διευθυντής Κέντρου Μελετών, Περιφερειακών Μελετών, στο Γερεβάν της Αρμενίας. Επίσης, καλωσορίζω την παρουσία του πρεσβευτού της, Ευρωπαϊκής, ε, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστού μας, γνώριμου μας, του πρεσβευτού Γένελ. Και επίσης δεν ξέρω αν έχουμε εδώ τον ε, πρεσβευτή της Αρμενίας, όχι ή τον ε, πρώτο σύμβουλο της ε, πρεσβείας, ο οποίος ασφαλώς είναι εδώ σας καλωσορίζω και είμαι βεβαία ότι θα έχετε την ευκαιρία και να ε, τοποθετηθείτε Η ιδέα λοιπόν είναι το πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να συμβάλλει σε μια διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας επί τη βάση δεσμεύσεων του 2009 που ξεκίνησε με τα πρωτόκολλα το 2009, που τα οποία όμως εντωμεταξύ δεν έχουν επικυρωθεί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη χώρα. Και έτσι εμείς ως βουλευτές θα θέλαμε να δούμε τι είδου ε, πρωτοβουλίε θα μπορούσαμε να αναλάβουμε πέραν της παρούσης συνεδριάσεως για να συμβάλλουμε στην διαδικασία της ε, συμφιλίωσης, η οποία για μας σημαίνει ανάληψη των διπλωματικών σχέσεων, επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων και διευκόλυνση της κυκλοφορίας, της κινητικότητας πέραν των συνόρων. Για να αντιληφθούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση, σε ένα πλαίσιο περιφερειακό, σε δεδομένα στην περιφέρεια αυτή ε, πολύ διακειμενόμενα, πολύ ασταθή και αβέβαια, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Ασφαλώς θα μας μιλήσετε για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, αλλά δεν λησμονούμε και τις τελευταίες αποφάσεις ε, της Αρμενίας για ένταξη στην Τελωνιακή Ένωση σε ένα χώρο μάλιστα με τον οποίο δεν έχουν ουδέν ουδέν κοινό σύνορο, πράγμα το οποίο μας φαίνεται κάπως παράξενο, αλλά και του θέματος των ενεργειακών πόρων, οι οποίοι ασφαλώς έχουν την ιδιαίτερη τους βαρύτητα στην υπόθεση αυτή. Ως οικολόγος έχω τις απόψεις μου, ασφαλώς δεν είμαι η μόνη η οποία κρίνει έτσι τη σημασία των ενεργειακών πόρων στις διεθνείς σχέσεις. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνδιοργανωτή και πρόεδρο, συμπρόεδρο εδώ, τον κύριο Σάμπανοτς, το φίλο Μίλαν. Μου επιτρέψει να σε λέω Μίλαν για να απλουστεύουμε τα πράγματα. Να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα με το όνομα. Μίλαν είναι το δικό μου όνομα. Τσαμπερνόχ είναι το οικογενειακό όνομα και είναι πολύ δύσκολο πρόφερτο για πολλούς ξένους. Με τα χαρά σας υποδέχομαι όλους. Εκτιμώ την ύπαρξη αυτής της σα Ασυνήθη σύνθεση. Ε, ίσως έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. Εκτιμώ που έγινε αυτή η συνδιαργάνωση των, με τις δύο αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με μια αρμόδια επιτροπή. Χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω τους ε, ομιλητές μας. Να επενθυμίσω ότι στα πλαίσια της τελευταίας συνεδριάς Επιτροπής με την Εθνοσυνέλευση Αρμενίας στην Επιτροπή Συνεργασίας, πέρσι τον Νοέμβριο στις ε, το, στις Βρυξέλλες. Καταγγείλαμε ότι τα πρωτόκολλα δεν έχουν επικυρωθεί ακόμα. Θέλαμε ίσως να βρούμε και κάποια εναλλακτικά πρωτόκολλα για να πετυχαίνουν τους ίδιους στόχους ή να επικυρωθούν αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας. Ε, με τα χαράς δέχομαι και τα παρόντα μέλη, τους εμπειρογνώμονες που θα ασχοληθούν με τα εξής Πρώτα απ' όλα, πως η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας της Αρμενίας ε, που θα ε, είναι το 2015 επηρεάζει τις προπτικές για τη διοργάνωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών ε, των πολιτικών Αρμενίας και Τουρκίας στον τομέα αυτό. Θα μπορούσαν να απτυχθούν προγράμματα εντατικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους τους διεθνείς φορείς όσον αφορά τον οικονομικό και πολιτικό τομέα, ώστε να πιστούν οι δύο χώρες να επαναλάβουν τις συνομιλίες όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ε, σχετικά με αυτό λοιπόν, μας ε, είπαν οι αρμόδιοι φορείς ότι το μέσο για τη σταθερότητα θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των προσπαθειών των διπλωματικών στη δεύτερη φάση μεταξύ των δύο χωρών. Η εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μας ε, ενημερώσει σχετικά με αυτό και πώς οι εσωτερικές πολιτικές δυναμικές στην Αρμενία και την Τουρκία επηρεάζουν την δυνατότητα εξομάλυνσης των ε, σχέσεων. Ε, είναι ε, οι συνέπειες της μεταρρύθμισης του συντάγματος και πώς επηρεάζει και η επίλυση του κουρδικού προβλήματος στην Τουρκία την όλη κατάσταση και τι, επίσης και τι γίνεται και με το πρόβλημα της επανένωσης της ε, Κύπρου. Ε, ενδιαφέρει τα μέλη πώς εμείς σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ε, τι περιμένετε εσείς από εμά. Είναι κρίσιμο. Απλό ερώτημα αλλά κρίσιμο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Τι μπορούμε να κάνουμε μετά τις εκλογές ή τι μπορούν να κάνουν οι συνάδελφοί μας ε, της επόμενης αιτίας, την επόμενη πενταετία. Διότι δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν πετύχαμε πολλά το, την προηγούμενη πενταετία και θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ε, θα καλέσω τώρα τους φιλοξενούμενους μας να κάνουν τις παρουσιάσεις τους, τους εμπειρογνώμων. Τον καθηγητή Τζέγκη Αχτάρ και τον κύριο Ρίτσαρτ Γκεργοσιάν. Οι οποίοι έχουν το λόγο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μέραμπα, αρενσές ή Αξαμλάρ. Θα μιλήσω αγγλικά, αλλά μετά θα γυρίσω στα γαλλικά και ίσως και στα τουρκικά. Για να κάνω το φίλο Κερέμ που βρίσκεται στην ε, τουρκική καμπίνα, παλαιό φίλο και διερμηνέα, να δουλέψει. Θα περίμενε να, δουλέψω, να μιλήσω γαλλικά, αλλά εγώ θα μιλήσω αγγλικά πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, Σέμπερνότς, κύριε Πρόεδρε Σέμπερνότς, τα είπα σωστά. Ελένα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που αναλάβατε την πρωτοβουλία για το θέμα της, των σχέσεων Τουρκίας και Αρμενίας. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν απασχολεί την καθημερινότητα, δεν είναι αυτονόητο στην θεματολογία του σεπτού αυτού ακροατηρίου. Η Ελέν με πρόλαβε με το λάψους της ε, μιλώντας για τουρκο-ευρωπαϊκές σχέσεις αντί για τουρκο ερμενικες αλλά μου άρεσε αυτό το λάψους, ήταν χαριτωμένο και χαρακτηριστικό. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα ήθελα να σας ε, παραπέμψω στην έκθεση που καταρτήσαμε για το Κοινοβούλιο που καταγράφει τις θέσεις μας και να πω προφορικά κάποιες ιδέες για την μοίρα των πρωτοκόλων του 2009, ε, τα οποία τα περιγράφω στο έγγραφο, στην έκθεσή μου, ως ε, παγωμένα έως θανάτου ή ιδάλως λησμονημένα 100% στη χώρα μου τουλάχιστον, την Τουρκία. Η ενεργητικότητα του Υπουργείου Εξωτερικών της ε, Τουρκίας αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στη Συρία και ίσως και λίγο στην Αίγυπτο, αλλά δεν ε, αφιερώνονται πόροι και ενεργητικότητα σε θέματα όπως αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρο Τσάμπερνο, όπως την Κύπρο ή τις σχέσεις με την Ελλάδα ή ακόμα και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σχέσεις λοιπόν με την Αρμενία και η εξομάλυνσή τους έχουν και αυτές πολύ, λίγη, πολύ λίγο μερίδιο της προσοχής του Υπουργείου Εξωτερικών και του προσωπικού του. Και άρα θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος. Υπάρχει τρόπος να αναζωογονηθούν τα πρωτόκολλα, κάποια ε, διάθεση φαίνεται να διαγράφεται από τον έντιμο με διαμεσολαβητή όπως ονομάζεται Honest Broker, την Ελβετία δηλαδή, για επαναφορά του θεματολογίου τόσο στο Γερεβάν όσο και στην Άγκυρα και βέβαια και την Κωνσταντινούπολη έχουν αποδειθεί σε προσπάθειες διαμεσολάβησης. Τι μπορούμε ε, λοιπόν να σημειώσουμε ως προς το θέμα αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται non-issue, σαν ανύπαρκτο δηλαδή αυτή την εποχή. Όσον αφορά την Τουρκία, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο παράγοντες. Καταρχάς τον παράγοντα Αζερβαϊτζάν, ο οποίος μπορεί να ήταν λιγότερο ορατός ή καθοριστικός στην κατάρρευση των, των πρωτοκόλων, ε, κατέστησε το χρόνο στρατηγικής σημασίας παράγων και καθορίζει σήμερα την ε, πολιτική της Τουρκίας έναντι της Αρμενίας και ακόμη έναντι των Αρμενίων εν γέννη. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο ο Ρίτσαρτ βλέπω ότι συμφωνεί μαζί μου. Είναι ένα νέο στοιχείο λοιπόν και πρέπει να το έχουμε υπόψη. Η έποψη των Αζερίων είναι ξεκάθαρη. Δεν θα πρέπει η Τουρκία να επιτραπεί να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Αρμενία, εκτός και αν η Αρμενία επιστρέψει το Ναγκόρνο Καραμπάχ Κάτι το οποίο βέβαια απαιτεί πολλές απαντήσεις, αφήνει πολλές ε, φαιές ζώνες και πάντως ε, όσο και αν δεν είναι τόσο σαφής και περίφραση τοποθέτηση των Αζερίων είναι ξεκάθαρη. Και έτσι θα πρέπει να ε, εδρεωθεί η θέση της Τουρκίας ως προς το ζήτημα του Καραμπάχ κατά την εποχή των πρωτοκόλων. Το Αζερβαϊτζάν είχε μια ενεργό στάση στην υπόθεση αυτή, αλλά εντωμεταξύ έχει αναπτύξει μια πολυεπίπεδη στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Και λαμβανωμένη υπόψη ε, της όλο και διεγκούμενης ανάγκης που έχει η Τουρκία σε περισσότερους ενεργειακούς ε, πόρους, έχει πιέσει στον τομέα αυτών. Η ΤΑΝΑΠ, η διανατολική ε, αγωγή, Trans-Anatolian Pipeline, έχει υποκαταστήσει το πρόγραμμα για τον Αμπούκο. Η ΣΟΚΑΡ η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερβαϊτζάν έχει μεγάλο μερίδιο από την Πέτκιν, την, ε, τον, κολοσσό, τον πετρελαϊκό κολοσσό της Τουρκίας και ο πρόεδρος της, Αζέρος, δήλωσε πρόσφατα ότι και η Σόκαρ και το Αζερβαϊτζάν εν γέννη ήθελαν ε, να γίνει τεράστια επένδυση έως το 2017, 17 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία. Να γίνει ο μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας για το πετρέλαιο του Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν συμμετέχει σε άλλες, σε κοινοπραξίες ε, με τουρκικούς ομίλους, εξαγοράζει ε, από τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες μέχρι τα πάντα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση στην αγορά της Τουρκίας. Αυτή η εταιρική, στρατηγική η εταιρική σχέση δεν πάβει όμως σε αυτά. Το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία έχουν πολύ στενή συνεργασία στο ευαίσθητο θέμα του, της γενοκτομίας και κυρίως εν ώψη της 100ης επαιτίου του 2015. Αντίστοιχα υπάρχει μια διαδικασία ευαισθητοποίησης, μια εξαρτή ευαισθητοποίησης για το ζήτημα του Καραμπάχ στην Τουρκία και πολύ στενή παρακολούθηση ασδήποτε δραστηριότητας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, Τουρκία και Αρμενίας δηλαδή, και παραμένουν αυτές στο στρόχαστρο του Αζερβαϊτζάν, το οποίο διατηρεί γενικό προξενείο στο Κάρς της Τουρκίας, πολύ κοντά στα αρμενικά σύνορα, και θα ήθελα να σας δώσω την εξή πληροφορία τις εξή πληροφορίε, Μια αναφορά πριν από 2-3 χρόνια περίπου, την οποία είχαν αναλάβει ως πρωτοβουλία οι ίδιοι οι κάτοικοι του ΚΑΡΣ, της πόλης του ΚΑΡΣ, ζητώντας να ανοίξουν τα χερσαία σύνορα, στην οποία απάντησε με, μια επιθετική, με ένα επιθετικό διάβημα το προξενείο, το αρζερικό προξενείο στο ΚΑΡΣ, ε, χρησιμοποιώντας άρθρα και δημοσιεύσει εφημερίδες για να καταρρύψει τέτοιου είδους επιχειρήματα και ε, αυτή την εκστρατεία των πολιτών του ΚΑΡΣ. Και μια δεύτερη πρωτοβουλία, ένας ιδιώτης επιχειρηματίας αποφάσισε να να οργανώσει μια αεροπορική διαδρομή μεταξύ του, του Βαν της Τουρκίας και του Γερεβάν της Αρμενίας. Μέχρι τελευταία στιγμή πρόκειται να ξεκινήσουν οι πτήσεις, αλλά δυστυχώς την τελευταία στιγμή ματαιώθηκαν λόγω των πάρα πολύ σοβαρών πιέσεων των αζερικών αρχών στην Τουρκία, προξενικών αρχών. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι άλλο εν ώψη του ζητήματος ε, της μοίρα που μπορεί να έχουν στο μέλλον αυτά τα πρωτόκολλα. Και αυτό έχει να κάνει με, τις, ε, με την εσωτερική διελκυστήριντα και τις συνθήκες στην εσωτερική πολιτική ζωή της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένα, ένα εκλογικό μαραθώνιο, γιατί έχουμε πρώτα δημοτικές εκλογές, ακολουθούν προεδρικές εκλογές και στη συνέχεια γενικές εκλογές, που θα μας πάνε μέχρι τα μέσα του 2015. και οι οποίες προφανώς περιορίζουν τις ε, δυνατότητες χειρισμών και κινήσεων τόσο της κυβέρνησης όσο και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ενδεχομένως με τη μορφή παραχωρήσεων σε θέματα ευαίσθητα όπως σε σχέση με την Αρμενία. Αλλά όχι μόνο εκεί, σας αναφερθήκατε στο κουρδικό ζήτημα, το ίδιο ισχύει και εκεί. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι υποχωρεί, ότι παρετείται έναντι ασδήποτε πιέσωση και στόχου που θα οδηγούσαν σε μια πιο φιλελεύθερη πολιτική μέσα στη χώρα. Άρα, και αυτό με το φόβο ότι μπορεί η εθνικιστική κοινή γνώμη να αισθανθεί ε, προσβεβλημένη και ως εκ τούτου να ε, εγκαταλείψει την υποστήριξη, να ε, πάψει να υποστηρίζει το κυβερνόν κόμμα. Μπορεί να είναι εσφαλμένη αυτή η εντύπωση, αλλά πάντως αυτή είναι η εντύπωση που έχει το κυβερνών κόμμα. Πριν ακόμη από το θέμα της ε, Αρμενίας. Τα θέματα αυτά ήταν ένα από τα σοβαρότερα ε, προσκόμματα στην επίλυση των διαφορών με τους Κούρδους. Τώρα, μία λύση, μία εξαίρεση σε όλο αυτό το πλέγμα σχέσεων και τοποθετήσεων θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος Γκουλ Ξέρετε ότι υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία με την διπλωματία του ποδοσφαίρου. Το 2010 επισκέφθη σε ποδοσφαιρικό αγώνα το Γερεβάν, μεγάλη πρεμιέρα θα λέγαμε, μια πρώτη επίσκεψη στην ιστορία Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Αρμενία, ο οποίος μάλιστα είχε εκδηλώσει και ε, λύπη για την αποτυχία της ε, διαδικασίας εξομάλυνσης. Συμβολική σημασία χωρίς περαιτέρω. Στο Επίσημο πεδίο, αυτά έχουμε, αυτά είναι τα δεδομένα, περισσότερα δεν διαθέτουμε, αλλά πολλά άλλα πράγματα είναι ε, εν εξελίξη στην κοινωνία των πολιτών και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην Αρμενία θα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. γιατί εκδηλώνεται μια υποστήριξη, μια αλληλεπίδραση πάρα πολύ ισχυρή μεταξύ των δύο κοινωνιών, με συμμετοχή όλο και περισσότερο της ομογένειας και ασφαλώς πολύ σημαντικό είναι το ότι πλέον πάβει να είναι ταμπού το ζήτημα της ιστορικής μνήμης ή της ε, ιστορικής αμνησίας σε σχέση με το αρμενικό ζήτημα. Αυτό καταγράφεται και αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικούς ε, πυλώνες που έχω καταγράψει στην έκθεσή μου στο έντυπο που έχετε. Ίσως χρειαστώ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα ήθελα για να σας τα ε, εκθέσω, αλλά ίσως να δοθεί ευκαιρία. Καταρχάς, επικοινωνία μεταξύ των ε, πανεπιστημιακών ερευνητών κτλ. και γενικά δημοσιεύσει, γιατί όλο και περισσότερα είναι τα βιβλία για την ε, Αρμενία, τους Αρμενίους, την ιστορική αλήθεια, τι συνέβη, τι πραγματικά συνέβη στην Αρμενία με τους Αρμενίους. Όλα αυτά λοιπόν δημοσιεύονται συνέχεια στην ε, Τουρκία και είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, μια διαρκώς εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη διαδικασία ε, ευαισθητοποίησης, γνώσης που ε, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Επίσης έχουμε έρευνα στην ιστορική μνήμη, ατομική αλλά και συλλογική. Όλο και πιο πολλοί είναι οι Τούρκοι που ανακαλύπτουν ότι είναι αρμενικής καταγωγής ή ότι έχουν συγγενείς αρμενικής καταγωγής, πράγμα το οποίο στο παρελθόν αποτελούσε ταμπού και αποτελεί μια διαδικασία που όλο εξελίσσεται και γιγαντώνεται. Ε, βλέπουμε πολλούς Τούρκους που ζητούν τώρα να βαπτιστούν επειδή έχουν ρίζες αρμενικές. Μπορεί αυτό να μην γίνεται κάθε μέρα αλλά ήταν αδιανόητο πριν από λίγο καιρό. Τέταρτον, η α, συνείδηση και η ορατότητα των θεμάτων αυτών και πρέπει να πω ότι πριν από την δολοφονία του καλού μου φίλου Χραντ, του οποίου τη μνήμη τιμώ εδώ σήμερα, ήταν πολύ πιο περιορισμένη η ορατότητα των Αρμενίων. Οι μη μουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρκία δεν είχαν ορατότητα, δεν ήταν ορατές στο παρελθόν. Τώρα όμως είναι όλο και πιο παρούσες είναι όλο και πιο ε, έντονη η διεκδίκηση του ότι είναι Φερρυπίν Αρμένοι, διεκδικούν τη διαφορά τους, το ίδιο ισχύει όμως και για τους Ρουμ, όπως τους με τους Ρωμιούς, Έλληνες, αλλά και για τους ε, Εβραίους και ούτω καθεξής. Ε, επίσης, η θρησκευτική τοποθέτηση, όταν μιλάμε για ταμπού που εγκαταλείπονται και για ιστορική μνήμη, αυτή η ιστορική μνήμη. Δεν σημαίνει απλώς ότι αναζητούμε τις κακές, τα κακά γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα στο παρελθόν μας. Έχουμε μειονοτικές ομάδε Τουρκία, οι οποίες υπήρξαν στην ιστορία μας, έχουν παραγάγει και έχουν παραγάγει όχι μόνο αγαθά, αλλά και πολιτισμό και κουλτούρα. Πράγμα το οποίο επίσης καθημερινά ανακαλύπτει ο Τούρκος πολίτης και αποτελεί μια πολύ θετική και υγιή εξέλιξη. Και μια τελευταία λέξη θα πρέπει πιστεύω εδώ να αναγνωρίσουμε το out Caesar, out nihil. Είτε ε, ο Κέσσερ είτε τίποτα, δηλαδή ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση μη τι άλλο αυτές τις πρωτοβουλίες που οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις τα τελευταία δέκα χρόνια. Κάτι το οποίο δεν ήταν καν δια, ε, νοητό πριν από δέκα χρόνια, έστω και αν δεν ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτές τις εξελίξεις, ναι ίσως εν μέρη, η αναστήλωση της μεγάλης εκκλησίας στο Βαν, της εκκλησίας του Αχταμάρ, ε, ήταν ένα σημαντικό γεγονός ε, ή μη τι άλλο δεν ε, ε παρεμποδίζει τέτοιου είδου πρωτοβουλίες η κυβέρνηση και αυτό πάλι θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Και να το σημειώσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι μπορώ να ολοκληρώνω, ίσως ένα δύο λεπτά ακόμα. Το κοινοβούλιο λοιπόν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά όχι μόνο αυτά, και τα αμερικανικά, γενικά η Δύση. Καλό θα ήταν να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Εσείς, Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο μέσο σταθερότητας που δρομολογείται και εμείς έχουμε μπλεκεί με τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Τουρκία και άλλες τέσσερις από την Αρμενία που θα συνεργαστούν, οι οποίες ήδη συνεργάζονταν, όμως με την στήριξη τώρα των ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορούμε να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε ίσως και τα όσα γίνονταν από τις 8 αυτές με κυβερνητικές οργανώσεις. Πολλές πρωτοβουλίες την χάνουν υποστήριξης και διμερός από τους Γάλλους Φερπίνη, από τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς και ασφαλώς και από την τουρκική κυβέρνηση. Η έκθεση στην οποία αναφέρεται η Ελένα στο ισόγειο επί παραδείγματι την χάνει υποστήριξη είναι υπό την αιγίδα της Βρετανικής και της Ολλανδικής κυβέρνησης. Και έτσι μπορούμε νομίζω να πούμε ότι προχωρούμε προς μια εξομάλυνση, μπορούμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη, μια εξομάλυνση η οποία θα αναπτυχθεί πάνω στις ε, πρωτοβουλίες αλλά και θα προκαλέσει πρωτοβουλίες ε, των δύο κυβερνήσεων. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ακτάρ για την παρουσίαση αυτή που μας καλεί να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. Να, ένα καλό μήνυμα. Ο κύριος Κυραγκοζιάν, έχετε ετοιμάσει ε, μια σχετική έκθεση με την οπτική γωνία από την άλλη μεριά των συνόρων. Ε, για πείτε μας λοιπόν μερικά πράγματα για πρωτοβουλίες που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Πρώτα πρώτα να σας αναφέρω το ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί πιστεύουμε ότι το ζήτημα δεν υπέραν πέραν της Τουρκίας και της Αρμενίας. Υπάρχουν δύο παράμετροι που κάνουν το θέμα επίκαιρο. Πρώτον, σε, στην ευρύτερη περιφερειακή περιοχή η Αρμενία είναι η μόνη περιοχή η οποία είναι σημαντική για το μέλλον στο Νότιο Κάφκασο θα έλεγα μετά από τα τελευταία πέντε χρόνια τον πόλεμο Τουρκίας-Γεωργίας οι σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να ε, έχει μια κάποια αισιοδοξία η προσπάθεια λοιπόν των καλών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας είναι σημαντική είναι μια κοινή προσπάθεια και προσπαθούμε να πούμε και στις δύο κυβερνήσεις ότι εκείνο που είναι σημαντικό είναι να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση. Δεν πρόκειται για προπαγάνδα, δεν πρόκειται για εφεύρεση αφηγημάτων σχετικά με το τι συμβαίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε προς το μέλλον, όχι να είμαστε όμοιροι του παρελθόντος. Ας αρχίσω όμως για τα, από τα πρωτόκολλα. Η υπογραφή των πρωτοκόλων αυτών καθεαυτών μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας απαιτούν επιτυχία στην ε, συνιστούν επιτυχία στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη τα πρωτόκολλα. Αλλά οι αμοιβέ επισκέψεις των αρχηγών κρατών που πήγαν από τη μια χώρα στην άλλη ήδη ήταν ένα βήμα μπροστά και ήταν επιτυχία. Επίσης, ακόμη και αν τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας παραμένουν κλειστά, έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα πνεύματα, να ανοίγουν τα μυαλά και από τη μια και από την άλλη μεριά. Και αυτό είναι πρόοδος. Επίσης, αν δούμε τι, ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζεται, τα πρωτόκολλα στη τελευταία ανάλυση είναι πολύ πιο σημαντικά για αυτά που δεν λένε από ό,τι για αυτά που λένε. Τα πρωτόκολλα δεν αναφέρονται καθόλου ούτε ακροθυγός και δεν αναφέρουν καθόλου ούτε τον Αγκόρνο Καραμπάχ ούτε την αρμενική τη γενοκτονία των Αρμενίων τα πρωτόκολλα αυτά καθε αυτά είναι ουσιαστικά μια διόρθωση της πολιτικής γιατί με την έννοια ότι η Τουρκία καλείται να διορθώσει και να αλλάξει πολιτική το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι φυσιολογική δράση στα πλαίσια μιας εξωτερικής πολιτικής και σίγουρα δεν ήταν και παραγωγική κίνηση τα πρωτόκολλα επίσης είναι πεπαλαιωμένα ήδη άμα λάβει κανείς υπόψη ότι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο κάνουμε τώρα είναι ότι εφαρμόζουμε τις, τις πιο μετριοπαθείς ρήτρε των πρωτοκόλων να υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις ενδεχομένως να ανοίξουν τα σύνορα αλλά εδώ πρόκειται όμως για διαδικασία εξομάλυνσης όχι συμφιλίωσης η συμφιλίωση είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία και πολύ πιο μακροπρόθεσμη. Η εξομάλυνση όμως είναι το πρώτο βασικό προαπαιτούμενο για τη συμφιλίωση. Δηλαδή το να ανοίξουν τα σύνορα και να υπάρχουν δημοκρα... διπλωματικές σχέσεις είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνεται σήμερα. Είναι το πρώτο βήμα θέλετε για τη συμφιλίωση μπορεί. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι το εξής. Πού βρισκόμαστε τώρα Πρώτα πρώτα είμαστε όμοιροι της εσωτερικής, της εγχώριας πολιτικής στην Τουρκία και ο πραγματικός κίνδυνος είναι να διαρκέσει η διαδικασία ή η αναστολή ή το πάγωμα των διαδικασιών τόσο πολύ ούτως ώστε η Τουρκία να αρχίσει να είναι μη ειλικρινής ως συνομιλητής και όσο περισσότερο περμένουμε τόσο πιο ρεαλιστικό θα είναι να πούμε ότι θα χάσουν την υπομονή τους οι Αρμένοι. Συγχρόνως υπάρχουν σημαντικά επιτεύγματα ε, όσον αφορά την έλλειψη αν θέλετε προϋποθέσεων δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα από καμιά πλευρά και αυτό συνεχίζεται. Άμα δούμε το ρόλο τώρα κάποιων εξωτερικών παραγόντων, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ρωσία παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να επεκτείνει την εξουσία της προς τον Νότιο Κάφκασο, η Ρωσία επέτρεψε στη διαδικασία αυτή εξομάλυνης Τουρκίας-Αρμενίας να εξελιχθεί. Και η Δύση, εγώ σαν Αμερικανό-Αρμένιος λέω, ιδιαίτερα οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Αυτό είναι καλό. Και τα πράγματα είναι πιο πραγματικά έτσι. Η Τουρκία πρέπει να επανυπολογίσει την πολι... και να διορθώσει την πολιτική της και δεν πρόκειται για μια Πρόκειται να γίνει μια κάποια ε, πρέπει να κάνει η Τουρκία μια ειλικρινή διόρθωση και όχι πράγματα ή έργα βιτρίνας για να ευχαριστήσει τη, Δύση τους Αμερικάνους. Τώρα το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικός παράγοντας για την τουρκική πολιτική αλλά και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ε, θυμώνεται θυμώνει από το γεγονός ότι το Αζερβαϊτζάν ουσιαστικά επιβάλλει βέτο στο Νότιο Κάφκασο. Ποιος, ποιος ε, έδωσε το δικαίωμα στο Αζερβαϊτζάν να είναι τέτοιο είδους τεράστιο εμπόδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μέσου σταθερότητας επενδύει πολύ σε αυτό στην δημιουργία καλών σχέσεων Τουρκίας και Αρμενίας και αυτό είναι καλό. Τους τελευταίους μήνες δημιουργείται μια, ένα καινούριο πολιτικό πλαίσιο. Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πρωτοκόλου θεωρήσουμε ότι οι αστερισμοί ευθυγραμμίζονται τώρα τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες έχουμε δείγματα ότι η Τουρκία στη, ε, ε, διαταράσσεται ή χάνει τη συγκέντρωσή του στο θέμα αυτό και λόγω Συρίας αλλά και λόγω εσωτερικής κατάστασης βλέπουμε διαδηλώσεις στην Τουρκία βλέπουμε διαδηλώσεις εναντίον του Πρωθυπουργού της Τουρκίας και της μορφής με την οποία διοικεί ε, και εδώ η και η Αρμενία έκλεισε την πόρτα στην Ευρώπη. Για μένα είναι κακό αυτό που έκανε η Αρμενία, αλλά η Τουρκία δεν ε, κλειδώθηκε η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επελέγησαν άλλα εργαλεία τελωνιακή ένωση κτλ. κτλ. Η... Αυτά είναι καλά για την εξομάλυνση αλλά βλέπουμε τώρα εδώ να φτάνει η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρμενίων και αυτό επιβάλλει πίεση και ψυχολογική ε, πίεση στην Τουρκία και στην τουρκική κυβέρνηση και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και ως μέλος διασποράς και ως Αμερικανού που μένω τώρα στην Αρμενία εκείνο που είναι ενδιαφέρον για μένα είναι ότι είμαι, μέλ, είμαι μέλος της διασποράς αλλά είμαι ουσιαστικά και μέλος της τουρκικής διασποράς ο παππούς μου ήταν από το Λαζίκ Τούρκος λοιπόν τελικά τα γεγονότα του 1915 ε, δημιούργησαν ένα μεγάλο μέρος της διασποράς και από εδώ και από εκεί. Αλλά θα ήθελα να πάω λιγάκι παραπέρα και να τονίσω το μέρος εκείνο της κοινή μας έκθεσης το οποίο είναι οι συστάσεις, κοινέ συστάσεις. Οι συστάσεις είναι αρκετά ρεαλιστικές. Εγώ είμαι ο αισιόδοξο, ο συνάδελφος είναι ο απεσιόδοξος, είμαστε όμως αρκετά ρεαλιστές. Πατάμε στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή της εξομάλυνσης. Την ορμή να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο και κάλυψη πολιτική και για τις δύο κυβερνήσεις για να προχωρήσει η εξομάλυνση. Από την άλλη μεριά η συνεργασία της κοινωνία των πολιτών και από τις δυο πλευρές είναι σημαντικό και η κοινωνία των πολιτών είναι πιο πολύ η κοινωνία των πολιτών πραγματικά από ό,τι στο παρελθόν και έτσι μπορεί να επέλθει μια κάποια συμφωνία που πρακτική πολύ πιο σημαντική από την συμφωνία σε διπλωματικό χαρτί. Οι κοινωνίες λοιπόν των πολιτών προσεγγίζουν μια την άλλη. Κάτι άλλο Θέλουμε να διευρύνουμε την έννοια της εξομάλυνσης και στο υπόλοιπο κόσμο πέρα από την ιντελιγέντσια της Κωνσταντινούπολης ή της Μύρνης. Θέλουμε και στις διάφορες περιφέρειες και στην Ανατολική Τουρκία να συνειδητοποιήσει ο κόσμος την εξομάλυνση και στην Αρμενία γιατί και εκεί πρέπει να ανατραπούν και ταμπού και αφηγήματα του παρελθόντος. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε κάποιους φορείς αλλαγής, οικονομικούς, τουριστικούς, ανταλλαγές ε, πανεπιστημιακών, ερευνητών, φοιτητών, για να προετοιμάσουμε την κατάσταση για τη δημιουργία διπλωματικών σχέσεων να, δημιουργεί, να κάνουμε πιο επίσημες τις άτυπες διπλωματικές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν να ε, Παραδείγματο χάρη, η Αρμενία είναι ιδρυτικό μέλος της οργάνους για, τη βόρεια, για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, ε, υπάρχει το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχουν τέτοιου είδους διεθνείς οργανισμοί όπου οι χώρες μας πρέπει να έρθουν πιο κοντά και πρέπει να, προετοιμάσουμε και την κατάσταση για σήμερα, για την, το άνοιγμα των συνόρων, να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για την πυρηνική για την ασφάλεια, για την ασφάλεια στα σύνορα, για την υγεία στα υπουργεία τα αντίστοιχα και των δύο χωρών για να μπορούν να δράσουν μετά το άνοιγμα των σύνορων. Και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συνελεύσεων της Τουρκίας και της ε, Αρμενίας και μπορεί, να εμπλακεί και το Αζερβαϊτζάν αλλά πρέπει να γίνουν πράγματα για να, δια, να υιοθετηθούν μηχανισμοί και χώροι συνάντησης ε, εναλλακτικοί και καινούργοι και να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να συμβεί αυτό γιατί το, η σημασία της υπόθεσης αυτής δεν πέραν των ορίων της Τουρκίας και της Αρμενίας γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή ότι είναι το μόνο θετικό πράγμα που συμβαίνει στο Νότιο Κάφκασο και για τη σταθεροποίηση και για τη σταθεροποίηση των περιοχών έξω ε, έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα με ρωτήσετε τι αποτελέσματα έχω, τι συμπεράσματα έχω. Δεν έχω συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή απλώς διατηρούμε την ορμή που έχει δημιουργηθεί, το momentum που έχει δημιουργηθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και από τις δυο μεριές των κλειστών συνόρων εμείς σαν πολίτες και από τη μια και από την άλλη μεριά θέλουμε παραπάνω πράγματα, θέλουμε καλύτερη κατάσταση και για την καθημερινότητα αλλά και για και στρατηγικά, πιο μακροπρόθεσμα. Πράγματα που έλειπαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Yes. Yeah, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στην εξοχότητά του τον κύριο Πρεσβευτή, τον κύριο Σετμιρέλ. Κύριε Πρέσβη, αν έχετε κάποια σχόλια ή αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ευχαριστώ Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω και διοργάνω συνεδριάσεως. Πριν ξεκινήσω, θα ποτίσω φόρο τιμή στην κυρία Ντίνκ που είναι εδώ μαζί. Άκουσα τον κύριο Ακτάρ και τον κύριο Κυραγκοσιάν. Προσεκτικά διάβασα προσεκτικότατα την έκθεση, άκουσα προσεκτικότατα ε, την έκθεση και άκουσα την όλη αφήγηση τους. Ε, δύσκολο να προσθέσω σε αυτά που υπόθηκαν, όμως υπάρχουν κάποια σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ανεξάρτητα από αυτά που μας είπε ο κ. Ακτάρ, το πρωτόκολλο δεν είναι νεκρό, Ίσως να μην είναι ζωντανά τα πρωτόκολλα, αλλά δεν είναι και νεκρά. Ε, θέλουμε να τα προωθήσουμε. Πιστεύουμε ότι μια δικασία εξομάλυνσης είναι προς όφελος και των δύο χωρών και προς όφελος της ε, περιοχής. Το άνοιγμα των συνόρων είναι σημαντικό, είναι ουσιώδες. Έχουμε παράδειγμα μπροστά μας. Πολύ δύσκολες σχέσεις είχαμε με το Βόρειο Ιράκ επί δεκαετίες και τώρα έχουμε παράδειγμα ανοιχτών συνόρων με αυτή τη χώρα. Ε, είναι προς όφελός μας να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρατε. Η εσωτερική πολιτική. Τα Τζερμπαϊτζάν παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο. Σωστά το είπατε. Τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και τίποτα άλλο δεν αναφέρεται στα πρωτόκολλα, αλλά υπάρχει, είναι στο υπόβαθρο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Δεν θέλουμε πλήρη λύση στο ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, θέλουμε κάποια βήματα όμως. Αν γίνουν βήματα από την αρμενική πλευρά θα υπάρξει ανταπόκριση. Κυρίως όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Αυτό θέλουμε όσον αφορά τη διαδικασία εξομάλυνσης. Δεν είναι η επίλυση του ζητήματος του ίδιου του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τι κάνουμε τώρα, όσοι έχουν τα πράγματα. Θέλουμε μέτρα δημιουργίας εμπιστοσύνης κλίματος εμπιστοσύνης. Και εκεί κάποια πράγματα έχουν γίνει, αναφέρατε κάποια πράγματα, θέλουμε να συνεχίσουμε, έχουμε αυτή την πρόθεση, μπορώ να σα δώσω διάφορα παραδείγματα, αναφέρω κάποια, υπάρχει ολόκληρο κατάλογο που έχω μπροστά μου, δεν θα σα κουράσω όμω θα χρειάζεται τα θέματα. Χιλιάδε παράνομα διαμένοντε Αρμένοι στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία και τα παιδιά του πηγαίνουν σε μειονοτικά σχολεία. Όσον αφορά τι τηλεπικοινωνίε, μεταφορέ. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα καλύψουμε σε πολιτισμικά θέματα, ανακαίνιση εκκλησιών που αναφέρατε, ιδιοκτησίες που επιστρέφονται ή αποκαθίστανται. Υπάρχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν, η κοινωνία αλλάζει στην Τουρκία, αυτό είναι σίγουρο και όπως είπατε συζητούνται περισσότερα αυτά τα πράγματα ποτέ στην Τουρκία. Όχι μόνο τα θέματα της Αρμενίας αλλά και το Οθωμανικό μας παρελθόν. Ε, είναι ε, μια συνειδητοποίηση του παρελθόντος που είναι υγιής όσον αφορά την περιοχή και πιο πέρα. Και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το τέλος του ψυχρού πολέμου συνεπέφερε μια ζωτικότητα στην όλη διαδικασία. Θέσατε άμεσο ερώτημα, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι τώρα μας ε, φέρατε μαζί μας, ενώσατε, αυτό είναι ήδη θετικό αλλά και ο χρονισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε δικασία. Μπορέσαμε να ετοιμάσουμε τα πρωτόκολλα λόγω κάποιου χρονισμού. Πρέπει να περιμένουμε για την επόμενη δυνατότητα, την επόμενη στιγμή στο χρονοχώρο που μπορούμε να κινηθούμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε. Και εκεί που παίξει ρόλο το κοινοβούλιο, στι επαφέ μεταξύ ανθρώπων, να ετοιμάζουμε και άλλε παρόμοιε συνεδριάσει. Διάφορε ιδέε να ακούγονται, διάφοροι τομεί των λαών να ακούγονται να μην είναι μόνο θέμα διαδικασίας εξομάλυνσης σχέσεων λαών, αλλά, ε, ε, χωρών συγγνώμη, αλλά εξομάλυνση σχέσεων μεταξύ λαών. Υπάρχει καχυποψία, παραπληροφόρηση, παρεξηγήσει και από τις δύο πλευρές. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι να έχουμε περισσότερες επαφές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι πολύ επικοδομητικό σε αυτό και από τη στιγμή θα έχουμε τη σωστή δυνατότητα και είναι η σωστή στιγμή μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειάζεται να ετοιμάσουμε το έδαφος για να προχωρήσουμε. Αυτά είναι τα σχόλιά μου σχετικά με αυτά που ήδη εκτενώς αναφέρθηκαν. Είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλη δυνατότητα, διότι μιλάμε και με εξομάλυνση της ιστορίας. Ευχαριστώ. Thank you, And now I would like... Ευχαριστώ, εξοχότατε. Μπορούμε να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Και Α, συγγνώμη. Μισό λεπτό παρακαλώ. Jill Spotman, επικεφαλής της ομάδας για την Τουρκία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα σας καθυστερήσω. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το πάνελ και τους ε, ομιλητές που ήδη ανέφεραν τις απόψεις τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας δύο πολύ τετριμένα ίσως πράγματα να, πούμε, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, συμφωνίες σύνδεσης και με τις δύο χώρες και τώρα διαπραγματεύεται με την Τουρκία συμφωνία προσχώρησης άρα υπάρχουν αυτές οι επαφές και δεύτερο βεβαίως είναι και προς το συμφέρον της Τουρκίας και προς τη, το συμφέρον της Αρμενίας να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ τους το ίδιο είναι και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια επικεντρώσαμε την προσοχή μας στις αλλαγές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ε, προφανές αυτό, όμως υπάρχουν πολλά ανεπίλητα ζητήματα στην περιοχή μας. Το θέμα της Κύπρου θα ξαναρχίσει τον επόμενο μήνα οι διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να επιτύχουν και μακάρι να επιτευχθεί πρόεδρος εδώ πριν από το 2015 όπως και ο Τούρκος ε, πρέσβης και εγώ δεν πιστεύω ότι τα πρωτόκολλα είναι νεκρά ήταν ένα βήμα μπροστά για το 2009 όταν υπεγράφησαν και θέλουμε πραγματικά η εξομάλυνση αυτή να γίνει χωρίς όρους να προχωρήσει χωρίς όρους και οι δύο πλευρές να παραμείνουν, να συνεχίσουν προσπάθειές τους για την εξομάλυνση. Τώρα, για την κοινή γνώμη, η, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό ευχαρίστως να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την επαφή των δύο κοινωνιών πολιτών αν θέλετε να σας πω, να σας αναφέρω ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη ξεκινάει για, για την υπόθεση αυτή. Θέλουμε να υπάρχουν επαφές μεταξύ των ατόμων, θέλουμε να προωθήσουμε πολιτιστικές και ε, άλλες δραστηριότητες, θέλουμε ανταλλαγή πληροφοριών με εξισορροπημένο τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο έργο που θα προχωρήσει, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα ε, πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει που βασίζεται στην ε, που βασίζεται στην ε, γαλλογερμανική, σε ένα γαλλογερμανικό παράδειγμα. Πάντως η EIS είναι έτοιμη να βοηθήσει όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χατζηγεωργίου. Well, so was... Ευχαριστώ πολύ. Με τα χαράς άκουσα τις ε, ομιλίες των δικαιοκριμένων ε, προσκεκλημένων μας. Ε, μας έδωσαν πολύτροφη προσκέψη. Θέλω να σχολιάσω εν συντομία και θέλω να δω τις αντιδράσεις σας. Πιστεύω ότι η Τουρκία έχει το πρόβλημα που έχει οποιαδήποτε μεγάλη χώρα όταν αντιμετωπίζει προβλήματα στη γειτονιά της. πρέπει να αντιμετωπίσει το ίδιο μέγεθός της η Τουρκία. Θα πρέπει να επεξεργαστεί το μέγεθός της. Είναι δύσκολο μια πολύ μεγάλη χώρα να συμπεριφέρεται γρήγορα, να κινείται γρήγορα, αντιδά γρήγορα. Παρόλο που η Τουρκία πρέπει σήμερα αυτό να κάνει. Είναι σαν ένα μεγάλο πλοίο που δεν μπορεί να, να στρίψει εύκολα και πρέπει να κάνει πορεία μιλίων για να βρει έναν τρόπο να περάσει από εκεί πρέπει. Σήμερα όμως η Τουρκία χρειάζεται γρήγορες αντιδράσεις προς το μέλλον, γρήγορες κινήσεις. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω και νομίζω ότι ακόμα και οι Ευρωπαίοι φοβούνται το μέγεθος της Τουρκίας. Πρέπει λοιπόν αυτό να αντιμετωπίσουμε και οι Ευρωπαίοι και οι Τούρκοι. Δεύτερον, είστε μέλο, μέλη ομάδων προβληματισμού και φοβούμε ότι πρέπει να σας πω κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη και να το αντιμετωπίσετε. Είπατε ότι πρέπει να δούμε το μέλλον και να μην είμαστε φυλακισμένοι του παρελθόντος. Πολύ συχνά, συνήθως, αυτές οι ομάδες προβληματισμού είναι όμοιροι του μέλλοντος. δεν μπορείς να συνδεθείτε με το παρόν, το, το σημερινό κόσμο. Λέτε, αναφέρετε πράγματα που είναι όνειρο, αλλά το όνειρο πρέπει να το συνδέσετε με αυτά που συμβαίνουν τώρα, επιτόπου. Φοβούμε, αυτή είναι η άποψή μου, ότι είστε πιο θετικοί από ότι μας υπαγορεύει η πραγματικότητα, μας δείχνει η πραγματικότητα. Το τρίτο. πρέπει να πω κάποια λόγια για το θέμα της Κύπρου. Επειδή κάποιοι εδώ αναφέρθηκαν στο θέμα. Ναι, μπορεί να αντιμετωπίσουμε την επόμενη εβδομάδα μια νέα πρωτοβουλία. Δεν θέλω να πω τίποτα, διότι οι Κύπροι απογοητεύτηκαν τόσες φορές κατά το παρελθόν, περιμένοντας λύση. Λοιπόν, σήμερα όλοι πρέπει να είμαστε ήρεμοι και βέβαια πρωτίστως η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η διαδρομή ίσως μας οδηγήσει προς το μέλλον. Και ελπίζω ότι επιλύοντας αυτό θα δούμε να ανοίγει ο διάδρομος για την Τουρκία. Διάδρομος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, καλωσορίζω τη σύζυγο του Χαραντίκ. Της εύχομαι θάρρος και να συνεχίσει ε, την πάλη που έκανε ο σύζυγός της κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur Ευχαριστώ κύριε Χατζηγεωργιού. Όπως και ο πρέσβης της Τουρκίας, ο κ. Γιανέλε, έτσι μπορεί να μιλήσει και ο κ. Μπιγιάγκοφ της αντιπροσωπείας της Αρμενίας. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε πολύ για τα πρωτόκολλα. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω και την ιστορία πώς εμφανίστηκαν αυτά. Από πού προήρθαν. Εδώ και πέντε χρόνια περίπου η Αρμενία ανέλαβε μια πρωτοβουλία. Την εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει χωρίς κάποιες προϋποθέσεις. Στόχος η δημιουργία διπλωματικών σχέσεων και το άνοιγμα των κλειστών συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Όλοι οι παριστάμενοι κατανοούν πόσο επώδυνο και δύσκολο ήταν αυτό σαν διαδικασία και σαν απόφαση για τους Αρμενίους, για την αρμενική κυβέρνηση. Όμως μας καθοδήγησε η ισχυρή πεποίθηση ότι αυτό το βήμα θα βοηθήσει να γυρίσουμε αυτές τις τραγικές σελίδε της ιστορίας και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και την ευμάρεια για τους λαούς μας και για όλη την περιοχή. Αυτό που συνέβη έκτοτε ήταν το εξής. Η Τουρκία απλώς αρνήθηκε να επικυρώσει τα πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν στη Ζηρίχη τον Οκτώβριο του 2009 μετά από ένα χρόνο εντατικοτά των διαπραγματεύσεων. Ο λόγος γι' αυτό, για την άρνηση, ήταν διάφορες προϋποθέσεις ε, που ετέθησαν σαν ζήτημα και σταμάτησαν τη διαδικασία. Αυτή είναι μια σύντομη παραπομπή στη σύγχρονη αυτή ιστορία των πρωτοκόλων. Ευχαριστώ. Thank και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος σε όλους εσάς για ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο κύριε Κύριλο, δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ πρόεδρε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο καλεσμένους μας για τις παρουσιάσεις που έκαναν οι οποίες ήταν πολύ επαγγελματικές θα έλεγα και μας ε, έδωσαν μια καλή, πολύ καλή εικόνα της κατάστασης. Συμφωνώ πως αυτά τα πρωτόκολλα όντως ήταν ε, το μόνο θετικό φαινόμενο στην περιοχή αυτή. Αν πάμε όμως παραπέρα υπάρχει τον Αγκόρνο Καραμπάχ Εκεί η κατάσταση είναι παγωμένη εδώ και κάμποσα χρόνια παρόλο που θα μπορούσε να εκραγεί. Και δεν είμαι ε, εχθρός ε, των... Ε, και δεν είμαι αντίθετος προς κάποιες κινήσεις, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει για να ε, διευθετηθούν, διευθετηθεί η κατάσταση. Εκείνο που θα μπορούσα βέβαια να σκεφτώ προφανώς όλα τα θέματα αυτά αλληλοσυνδέονται ε, το άνοιγμα των συνόρων, η εξομάλυνση των σχέσεων δεν μπορεί να ε, γίνει αν δεν γίνει έστω και ένα μικρό βηματάκι στην επίλυση του ζητήματος των Αγκόρνου Καραμπάχ. και εκεί και η Ρωσία και η Τουρκία θα πρέπει να εμπλακούν και ενδεχομένως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έστω, έστω ότι επιτυχάνεται συμφωνία για ένα μικρό βηματάκι απόσυρσης από μια γειτονική περιοχή. με τις απαραίτητες εγγύησεις ασφάλειας διότι βεβαίω η αρμενική πλευρά είναι πάρα πολύ ε, διστακτική στο να κάνει ορισμένες κινήσεις δίχως να υπάρχει και ένα μικρό αντίτιμο δεν ξέρω σας είπα ότι και οι, ε, τις αυτές και τις ασφάλειες μπορεί και να τις ε, παράσχουν και οι Ρώσοι και, άλλοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τη κατάσταση στην Γεωργία, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να σπρώξει λίγο την αμαξοστοιχεία. Η Ρωσία βέβαια μπορεί να θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι είναι προς το συμφέρον της να διατηρήσει την κατάσταση ως έχει. Αλλά μακροπρόθεσμα θα ήταν υπέρ της Ρωσίας να άνοιγαν τα σύνορα Τουρκίας-Αρμενίας διότι ο διάδρομος αυτός ενδεχομένως να είναι για την Τουρκία πιο καλός, πιο θετικός. Θέλω να πω λοιπόν ότι άμα φέρουμε μαζί και άλλους παίκτες στο παιχνίδι και Ρωσία και ομάδα Μιζ Λέει τώρα ο πρέσβης πρέπει να βρούμε πιο ρεαλιστικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιοχής. Ωραία. Λοιπόν, ένας πρακτικός τρόπος θα ήταν αυτός να ενώσουμε, να φέρουμε κοντά περισσότερους μεγάλους παίκτες στο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Ίσως να συνεργαστούμε με τη Γαλλία και να αναλυφθούν πρωτοβουλίες α, και από άλλους παίκτες. Ε, θα ήθελα να ακούσω τι σκέφτεστε γι' αυτό. Και τώρα να θέσω δύο ερωτήματα. Όσον αφορά την, τη διασπορά των Αρμενίων, ποια είναι η αντίδραση μετά την απόφαση για την ένταξη στην Τελωνιακή Ένωση. Άλλη ερώτηση. Αεροδρόμιο Νταγκόρνο Καραμπάχ. Το ζήτημα αυτό επελήθη. Φαίνεται να επελήθη. Έχει τον Αγκόνο Καραμπάχ υπάρχουν σχέδια να γίνει και αυτό μέλος της Τελωνιακής Ένωσης. I'm very open, Thank you for the Σε ευχαριστώ πολύ, Ευγένη, για τις ερωτήσεις. Και χαίρομαι που έθιξε στο ζήτημα ενός πιο ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Καζάκ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ε, πρεσβευτή και τους δύο ομιλητές μας για τη γενική και ρεαλιστική επισκόπηση της καταστάσεως καθώς και για τις προβλέψεις για την τόσο επιθυμητή βελτίωση, η οποία φαίνεται όμως προς το παρόν απίθανη στο ορατό μέλλον. Όλοι πάντως με καλή διάθεση νομίζω θα αρκούσε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα βήματα, έστω και αν, και αναφέρθηκε και αυτό νωρίτερα, δεν περνάνε αυτά από ένα πρωτόκολλο που αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο τουλάχιστον από πλευράς Τουρκίας. Και θα μπορούσαμε κάποια στοιχεία του πρωτοκόλου αυτού, στοιχεία κλειδιά, να τα αξιοποιήσουμε για συζητήσεις μεταξύ των δύο εταίρων, ώστε να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να ε, κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε στην εξομάλυνση, τη συμφιλίωση μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, λαμβανομένων υπόψη βέβαια των ευαισθησιών και τις δύο πλευρές ως προς κάποια σημεία της ιστορίας. Εγώ ως βούλγαρος βουλευτής τουρκικής καταγωγής μπορώ να πω ότι η ιστορία μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας έχει και εκείνη σημειώσει σημαντικά προβλήματα στα τέλη της δεκαετίας του 80, του 1980, περί το 89, όταν η μεγάλη ε, έξοδο την ονομάζουμε από τη Βουλγαρία ε, που οργάνωσαν η, η εκδίωξη από τη Βουλγαρία 300.000 ε, Βουλγάρων τουρκική καταγωγή από την Βουλγαρία προ την Τουρκία οδήγησε σε μεγάλη ένταση τη σχέση των δύο χωρών. Αλλά μετά το τέλο του κομμουνιστικού καθεστώτο και την θεαματική αναστροφή στην στάση τη κεντρική κυβέρνηση τη Βουλγαρία εναντί της τουρκική μειονότητα, σημειώνεται σημαντική και γρήγορη βελτίωση τη θέση μεταξύ των δύο λαών. Δεν είναι λοιπόν τίποτε το αδύνατο ή το απίθανο στην ιστορία. Αρκεί να πράξουμε το σωστό τη σωστή στιγμή και ο καθένας από την πλευρά του. Και οι δύο πλευρές, θέλω να πω, έχουν δρόμο να διανύσουν για να συναντηθούν. Να συναντήσουν όλο τον άλλον. Και συμφωνώ με τόσο είπε ο κύριος ο Κυρίλοφ ως προς το ότι θα πρέπει ίσως χωρίς να θέτουμε προϋποθέσεις απαραίτητα, αλλά πάντως ε, η κάθε χώρα και οπωσδήποτε και η Ερμενία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει με τη στάση της στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με την πρωτοβουλία του Προέδρου Γκιουλ και που οδήγησε στην πρώτη αυτή προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων. Μίλησαν οι δύο ομιλητέ μα για τι ειλικρινεί ε, συζητήσει τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αρμενία ε, και το διάλογο για τα θέματα του ιστορικού παρελθόντος που θα πρέπει να συνεχιστεί και με συγκεκριμένε δράσει σε επίπεδο πολιτικό πλέον. Δεν μπορώ παρά να ε, συμμεριστώ κι εγώ την πεποίθηση ότι και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο στο πλαίσιο της μικτής μας κοινοβουλευτικής επιτροπής όσο και στο πλαίσιο της Euronest οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις πλατφόρμες αυτές διαλόγου για να βελτιώσουμε τις επαφές, των διάλογο μεταξύ Τουρκίας, Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι όταν άκουσα τους δύο διακεκριμένους μας ομιλητές, Ακούγοντά του, μάλλον δεν μπορούσα να μην σκεφτώ τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μου. Είμαι Ευρωβουλευτή από την Κύπρο, ζω εδώ. Με ενθαρρύνουν πολύ τα όσα είπατε, ότι η κοινωνία των πολιτών, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αρμενία, κινείται, κινούνται οι κοινωνίε των πολιτών προ μία προσέγγιση. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μου. Οι κοινωνίε των πολιτών πάντοτε βρισκόνται μπροστά από τις ε, κυβερνήσεις και τους πολιτικούς πράγμα το οποίο κρίνω και ενθαρρυντικό και ευπρόσδεκτο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Κύπρο. Θέλουμε να υπάρξουν οι δραστήριοι αυτοί οι παράγοντες αλλαγής. Έχουμε think tanks, ομάδες αναλογισμού, προγράμματα, κοινέ επιχειρήσεις, τα προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω σημαντικός όμως και ο παράγον χρόνος. Όπως ανέφερε και ο αξιότιμος πρεσβευτής, εξοχότατος πρεσβευτής της Τουρκίας. Και δυστυχώς ο χρόνος πετά κιλά. Εάν λοιπόν δεν υπάρξουν κυρώσεις εάν αν δεν υπάρξει κύρωση ε, σε μια κυβέρνηση ώστε να υποχρεωθεί να ε, δώσει ένα τέρμα στους ε, διαχωρισμούς και τις διαιρέσεις σε μια κοινωνία, το μόνο που θα γίνει να περνάνε τα χρόνια και, να, και θα παραμένουμε εθεροβάμονες και ονειροπόλοι. Και εγώ ονειροπολούς από την δική των 18 ετών ότι μια μέρα θα επανενωθεί η χώρα μου και θα είναι ελεύθερη από τον ε, τουρκικό στρατό. Είμαι 58 ετών τώρα. Παραμένω ίσως οραματίστρια, αλλά τα όνειρά μου δεν έχουν υλοποιηθεί και περιμένω μία λύση. Ευχαριστώ όλους ε, τους ομιλητές για τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις τους ότι ενθαρρύνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, αλλά δυστυχώς εάν δεν ε, ε τα πραγματικά προβλήματα, αν απλώς ταχώνουμε κάτω από το ε, χαλή, ε, εάν δεν υπάρξουν προϋποθέσεις την ώρα που συζητούν η τουρκική και η αρμενική κοινή ε, γνώμη για αυτή τη διαφορά από τις χωρίες τόσες δεκαετίες, αν δεν συστηθεί πραγματικά το έχει συμβεί στον Αγκόρνο Καραμπάχ ή τι έχει συμβεί με, το, με την αρμενική γενοκτονία, αλλά και το τι συνέβη στην Κύπρο το 1974, μια τουρκική εισβολή η οποία προς, προσχηματικά ήρθε για να προστατεύσει υποτεθέτιους ε, τουρκοκυπρίους και έχει μείνει εντωμεταξύ πάνω από 30 χρόνια, 40 χρόνια στο νησί αν λοιπόν δεν δώσουμε απαντήσει σε αυτό που, ζητούν, ε, αυτό που ζητάει η κοινωνία των πολιτών, τότε μόνο ονειροπόλους μπορούμε να, ονειροπολία μπορούμε να προσφέρουμε, ονειροπόληση μπορούμε να προσφέρουμε στις προσεχείς ε, γενναίες. Αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ότι ούτε η Ευρώπη μπορεί να μείνει ε, αμέτωχη και άπρακτη εν των όσων πρακτούν τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία απλώς συλλέχουν ψηφίσματα από το 1974 έως το 2013, ψηφίσματα τα οποία μπαίνουν σε ένα σιρτάρι και δεν έχουν ποτέ εφαρμοστεί. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πράξει το ίδιο πολλά ψηφίσματα, πολλές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποφάσεις, αλλά μπαίνουν σε ένα σιρτάρι και δεν εφαρμόζονται ποτέ. Και κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, αν δεν υπάρξει μηχανισμός για την εφαρμογή των ψηφισμάτων και την επιβολή κυρώσεων όταν εφαρμόζονται όταν εγκρίνονται ψηφίσματα αλλά συνέχεια δεν εφαρμόζονται, τότε και του χρόνου εδώ θα είμαστε και παραπέρα εδώ θα είμαστε, ως κάποιοι από εσά πάλι, ε, με ένα όραμα πολύ ωραίο, αλλά μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα οράματα της κοινωνίας των πολιτών και την πραγματικότητα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, αν η Τουρκία έχει την πολιτική βούληση, και εδώ τελειώνω, εμείς λέμε ότι όποιος θέλει μπορεί. Εάν ε, η Τουρκία θέλει να λύσει τα προβλήματα με την Αρμενία και με την Κύπρο, να βεβαίω υπάρχει λύση πολιτική. Εφαρμόστε το πρωτόκολλο το σχετικό με την Κύπρο, εφαρμόστε το πρωτόκολλο το σχετικό με την Αρμενία και τελεία και παύλα. Πιέστε να γίνει αυτό λοιπόν. Επιβάλλετε κυρώσει. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε κύριε Παπαδοπούλου. Περιγράψατε πολύ καλά την κατάσταση πιστεύω. Ο κύριος Βάγκελ είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε δεν αρκεί η διοργάνωση συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που ίσως είναι πολύ ενδιαφέρουσες και η σημερινή είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε πάρα πολύ καλή επιχειρηματολογία από τους ομιλητές μας. Ίσως να μην χάνουμε και το χρόνο μας Απλώς θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Απευθυνόμαστε στους δύο προσκεκλημένους. Γιατί δεν αναφέρατε καθόλου τη Ρωσία σε αυτά που είπατε. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία όχι μόνο λόγω της Συρίας τώρα είναι σε διπλωματική επίθεση, αλλά είναι πολύ σημαντικός παίκτη στην περιοχή Ρωσία. Και από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, ο Κάφκασος ήταν το πεδίο για τις κινήσεις της Ρωσίας, για τον επεκτατισμό της Ρωσίας. Και δεν άλλαξε. Μέχρι σήμερα. Όταν μιλάμε για την Αρμενία δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η Αρμενία έχει ρωσικά στρατεύματα στο έδαφος της. Και τα ρωσικά στρατεύματα έπαιξαν ρόλο την κατάκτηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και τα ρωσικά στρατεύματα επιβάλλουν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Διότι η Αρμενία δεν κατέχει μόνο τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και αρκετές περιοχές γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η συζήτησή μας θα παραλύσει αν δεν θέσουμε επιτάπητος όλα τα στοιχεία. Η Αρμενία είναι δύναμη κατοχής. Δεν είναι ευπρόσδεκτη. Καταδικάστηκε από όλους τους διεθνείς φορείς για την εισβολή στον Αγκόρνο Καραμπάχ και για την αμετακίνητη θέση της όσον αφορά τις λύσεις για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ξέρετε, μιλήσαμε την ομάδα του Μίνσκ ότι αυτή ασχολείται με το θέμα. Ήμουν πρέσβης των ΟΑΣΕ στη Βιέννη εδώ και 20 χρόνια. Και η ομάδα του Μίνσκ ξεκίνησε τότε και παρόλα αυτά δεν πέτυχε τίποτα άλλο εκτός από το να αποδείξει ότι υπάρχουν διπλωμάτες, επιδέξει διπλωμάτες, έντιμοι άνθρωποι, μέλη της ομάδας του Μίνσκ, αλλά η λύση δεν είναι στα χέρια τους είναι πρωτίστως πολιτικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο. Είναι ακόμα μία παγωμένη σύγκρουση που θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Μία από τις πολλές. Διότι αυτές οι διαμάχες οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να μετατραπούν σε πόλεμο. Δεν βοηθά για λόγους προπαγάνδας να παραθέτουμε κάποιες διακηρύξεις ε, πρωθυπουργών, υπουργών αμήνης που απειλούν ε, προς τους για την εσωτερική τους πολιτική αυτοί οι άνθρωποι και λένε ναι έχουμε τη δύναμη να λύσουμε το πρόβλημα, θα το λύσουμε με κάθε θυσία με κάθε μέσο κλπ. Αυτά όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν. Όσον αφορά το μεγάλο προπολογισμό για τον εξοπλισμό του Ατζερμπαϊτζάν, βέβαια χρειάζονται έναν προπολογισμό. Δεν το χρειάζεται η Αρμενία, αφού είναι εκεί τα ρωσικά στρατεύματα. Και εγώ θα επικρίνω την Αρμενία. Τι στο καλό κάνουν, μπαίνοντα, συμμετέχοντα, προσχωρώντα στην ζώνη ελευθέρων συναλλαγών της Ρωσίας. Καθιστούν αδύνατη την ύπαρξη συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξαν πόκερ, έπαιξαν χαρτιά με πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Με πολύ μεγάλες προπτικές για τη χώρα. Και δεν ξέρω τι θα κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο για τις μελλοντικές προπτικές της Αρμενίας για να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αρμενία. Προφανώς αυτοί επέλεξαν ε, διαφορετική επιλογή. Και εφόσον δεν υπάρχει Αμερικανός διπλωμάτης ή πολιτικός εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς. Είδα το βιογραφικό σας. Συμμετείχατε σε όλους τους Αμερικανικούς φορείς λήψεως αποφάσεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε γιατί διστάζουν τόσο πολύ να παίξουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε αφήνουν το Αζερμπαϊτζάν να στριμώχνεται μεταξύ νέου εμπεριαλισμού της Ρωσίας και πολύ επικίνδυνου επεκτατισμού των Ισλαμιστών του Ιράν δεν αντιπροσωπεύει σοβαρότατη απειλή για τα συμφέροντά μας, για την ασφάλειά μας, για τα δυτικά συμφέροντα όσον αφορά την ασφάλεια. Αρκεί απλώς να διαβάζουμε τις ειδήσει για κάποια ανόητα πράγματα που κάνουν καμιά φορά οι Ατζερμπαϊτζαϊνοί όπως την υπόθεση Ζαφάροφ και να αφήνουμε τα ζητήματα σοβαρά παράμερα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Έτσι να το αντιληφθείτε. Θα καταλήξω αποδεχόμενος την ιδέα που ακούστηκε να ξεκινήσουν από κάπου οι δύο χώρες. Από κάπου σημαίνει η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Κάποτε, κάποτε εδώ και δύο χρόνια, ήμουν σε συνεδρίαση οργανώσεως της κοινωνίας των πολιτών με νέους από το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Δεν πυροβόλησαν ένα τον άλλον, ήταν φιλικοί, μπόρεσαν να μιλήσουν με τον άλλον παρόλο που ήταν προσεκτικοί να μην εκτεθούν στα μέσα ενημέρωσης κλπ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θα έπρεπε να το υποστηρίξουν. Ίσως η νέα γενιά έχει κάτι να πει, δεν ξέρω. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βάικολτ. Τέλος, ο κύριος Πέτερλε έχει το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω. Αυτά που άκουσα εγώ σήμερα, εδώ σήμερα είναι αρκετά ενθαρρυντικά και ε, εν γενή θα μπορούσα να συμφωνήσω. Ξέρουμε πόσο λεπτό και ευαίσθητο είναι το ιστορικό των τουρκο αρμενικων σχέσεων. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να βασιστούμε στην ιστορία για να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις. Δεν ξέρω επίσης κατά πόσον πράγματι βελτίωση αυτών των διμερών θέσεων θα βελτιώσει την κατάσταση σε ολόκληρη την περιοχή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα μπρος με καλή βούληση και καλές χειρονομίες. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Με την άδειά σας θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ένα ερώτημα και μετά θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Ερώτηση. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η Αρμενία αρνείται να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο στη διαδικασία Μίνσκ. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα αρχίζει, όποιος θέλει αρχίζει. Ευχαριστώ Μίλαν πριν να δώσουμε στους καλεσμένους μας το λόγο για να απαντήσουν ερωτήσεις, να μας κάνουν σχόλια θα ήθελα να εκμεταλλευθώ την παρουσία του, ε, από την παρουσία του της ε, κυρίας που είναι επιρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών για το θέμα και να της δώσω τον λόγο. Το μικρόφωνο κλειστό. Ναι, ευχαριστώ. Επανέρχομαι από ένα ταξίδι, με πρόσφατες λοιπόν ε, εντυπώσεις. Θα ήθελα να πω ότι βρίσκω πολύ συγκινητική την παρουσία της Ρακέλ Ντίνκ το χώρο αυτόν και τις ε, υποβάλλω το σεβασμό μου. Αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στο, στη σχέση ή τον κόμπο του Καραμπάχ στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Και να ρωτήσω τους δύο εδώ αναλυτές εάν ή σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκοπεί το ζήτημα του Καραμπάχ από τη διαδικασία για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Αρμενίας. Μιλισμονούμε ότι βρίσκεται σε ομοιρία έναντι του Αζερβαϊτζάν τώρα η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας για το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα και κυρίω προηγούμενο πολύ προς τον ε, κύριο Γκυραγκοσιάν από τις πληροφορίε που έχετε. Ενδεχόμενη αποχώρηση έστω μερική από μία από τις επτά επαρχίες, όπως τα λέγαμε, των των κατεχομένων περιοχών του Καραμπάχ δεν θα μπορούσε να έχει μια κάποια θετική ε, επίδραση. μια και μιλάμε για βήμα το βήμα, για συγκεκριμένα βήματα έναντι μια σύγκρουσης η οποία είναι χαρακτηριστική και της ε, παρακαταθήκης του κομμουνιστικού, του σοβιεστικού παρελθόντος που οδήγησε σε τόσες, ε, που ονομάζονται, παγωμένες συγκρούσεις και που έχουν να κάνουν βέβαια και με την αυτοδιάθεση των λαών αφενός αλλά και από την εξίσου σημαντική αρχή του απαραβίαση των συνόρων των κρατών αφετέρου. Και έτσι έχοντας επισκεφθεί και την Αρμενία και έστω και πολύ σύντομα, αλλά πολύ πρόσφατα το Αζερβαϊτζάν, θέλω να σημειώσω το πόσο πολλωμένες είναι οι κοινωνίες ως προς τα θέματα αυτά, πόσο πόλωση εκδηλώνεται και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εάν Μέσω ή μάκρο πρόθεσμα βλέπετε κάποια αλλαγή καθεστώς για τον Αγκόρνο Καραμπάχ και κάτι άλλο για σε 9 Οκτωβρίου και την ημερομηνία της δεξαγωγής για τις προεδρικές εκλογές στο Αζερβαϊτζάν 9 Οκτωβρίου. Υπάρχει περίπτωση βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αντιπροσωπεία για τη σχέση με τον Νότιο Κάφκασο να διατυπώσουν ένα αίτημα, μια διεκδίκηση, μια απέτηση διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως ε, μία ε, προώθηση ή υποστήριξη μιας ε, συμφωνίας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα που ίσως να μην έχουν ληφθεί υπόψη, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά η, η κατάσταση από πλευράς του Αζερβαϊτζάν μπορεί να είναι πολύχρωμη μπορεί να μπορούσε να κατανεμηθεί σε διαφορετικέ θέσει, επόψει και τοποθετήσει από πλευρά του Αζερβαϊτζάν. Αλλά ίσω θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί. Με συγχωρείτε που κάνω τόσε πολλέ ερωτήσει και τόσο μπερδεμένε, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα μου δώσετε το λόγο. Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και αν χρειάζεται να δώσουμε για κάποια ιστορικά στοιχεία. Η κυρία Φλότρο, όχι, σας βλέπω πολύ δυνατή και στον αυτοσχεδιασμό. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κύριε Φλότρη, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω, βέβαια θα κρίνει η Ρακέλ ίδια, αλλά θα ήθελα να προτείνω αν θέλει να λάβει το λόγο η ίδια. Η Ρακέλη Ντίνκ. Θα μιλήσω τουρκικά. Δεν σκοπεύω να μιλήσω. Είχατε ρωτήσει και πριν να αρχίσει η συνεδρίαση, αλλά εγώ από εκεί που βρίσκομαι, από την Κωνσταντινούπολη, δεν σκοπεύω να μιλήσω, εν πάση περιπτώσει μου είπατε α μιλήσω, α ακουστεί και δική μου φωνή. Με συγχωρείτε λοιπόν, με μία-δύο φράσεις μόνο θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ιδέες. Από τα όσα ακούω λοιπόν, από τα όσα παρακολούθησα, διαπιστώνω ότι για να μπορέσει κανείς να αναλύσει μια κατάσταση πρέπει να την έχει ζήσει. Πρέπει να έχει ζήσει ως πολίτης μιας χώρας ω μια κατάσταση στην πραγματικότητα. Μόνο έτσι μπορεί να την αναλύσει την κατάσταση. Αυτά τα οποία έχω ζήσει εγώ τα γνωρίζετε φαντάζομαι, αν όχι όλοι περισσότεροι. Είμαι Αρμένια, αλλά υπήκος της Τουρκίας και αυτά που θα σας πω και για τον Τούρκο υπήκο ε, είναι ε, αναφέροντας ότι στην υπηκότητά μου αλλά και στην ιδιότητά μου ως Αρμένιας. θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον όρο Τουρκιέλη που σημαίνει υπήκος Τουρκίας, αλλά θα πω Τουρκάλα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ακουστεί κάπως αρνητική αυτή η διατύπωση. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ιδέα που θέλω να εκφράσω και έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να ανεπτυχθεί κατά τρόπον ώστε να διδάσκει τον σεβασμό προς τον έτερο, την ε, ανοχή, την διαλλακτικότητα προς το διαφορετικό. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Τα σχολεία λοιπόν, σε αυτά θέλω να αναφερθώ. Τα παιδιά των Αρμενίων στην Τουρκία πηγαίνουν σε σχολεία ε, μειονοτικά, τα οποία όμως ε, απλώς τα κάνουν ανεκτά και δεν τους δίνουν ούτε ένα φύλλο χαρτί στο τέλος, γιατί δεν είναι ε, αναγνωρισμένο το δίπλωμα το οποίο ε, παίρνουν τελειώνοντας τα σχολεία αυτά. Σας το λέω ως μαρτυρία, σας το λέω γιατί το γνωρίζω από προσωπικούς ε, από προσωπική εμπειρία δεν μπορούν να γραφτούν μετά στο πανεπιστήμιο τα παιδιά αυτά όταν έχουν τελειώσει τα μειονοτικά σχολεία. Όσον αφορά τις εργασίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, πολύ καλά το να μην ε, προβάλλει προσκόμματα η κυβέρνηση Τουρκίας, δεν έχω καμιά αντίρρηση, ωραίο μου φαίνεται, αλλά ας δώσει και μια υποστήριξη για να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα αυτή η εξέλιξη στη σχέση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή ήταν μια άλλη πρόταση που θέλω να αναφέρω. Για για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ε, επιστρέφει στις, στις μειονότητες, ε, στις κοινότητες της μειονοτικές η τουρκική κυβέρνηση, θα το πω λαϊκά, σταγόνα στον ωκεανό ούτε ε, ένα κλάσμα από την αξία των περιουσιών που έχουμε χάσει. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα πρέπει να κάνει η τουρκική κοινωνία, το τουρκικό κράτο για να αναπτυχθεί η δημοκρατία περισσότερο. Όλα αυτά τα λέω επειδή γνωρίζω την Τουρκία. Σε αυτό μπορώ να μιλήσω. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Α αφήσουμε τα λεγόμενα δικαιώματα λουξ, τα δικαιώματα πολυτελεία. Α μιλήσουμε για τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα άλλο πράγμα θέλω να σας πω, πέραν της υποστήριξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρακολουθείτε την εφημερίδα μας, την εφημερίδα Άγκος. Μπορείτε να ενημερωθείτε για πολλά πράγματα, παρακολουθώντας την, διαβάζοντάς την. Με συγχωρείτε και πάλι για την αδεξιότητα και ευχαριστώ πολύ. Euh, euh, ευχαριστώ, Ρακέλ. Είχαμε επισκεφτεί τα γραφεία τη εφημερίδα από την αντιπροσωπεία, ήσασταν παρούσα και το ξέρετε, από την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ενώσεω Τουρκία και το Ίδρυμα και την εφημερίδα επισκεφτόμαστε που κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά για την ανοχή, την αναγνώριση της διαφοράς και για, τους, για ε, την υπηκότητα και τους πολίτες. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στους καλεσμένους μας, στους δύο καλεσμένους μας. Οι παρουσιάσεις τους ε, δημιούργησαν πολλές σκέψεις. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει συναισθηματική επένδυση που έχει γίνει που συνδέεται με την ιστορία, τραγική ιστορία. Δεν είναι μόνο τραγική, είναι και όμορφη όμως ιστορία πολιτισμικής παραγωγής, δημιουργία σχέσεων. Οι λύσεις που προτείνεται είναι ρεαλιστικές. Πράγματι, είναι η ευρωπαϊκή μέθοδος, πρέπει να πω, η μέθοδος της γερμανο-γαλλικής συμφιλίωσης που υποστηρίθηκε και αφέστηκε από τον Ζιλ Πόρτμαν θα ήθελα ενδεχομένω πάνω σε αυτό να επανέλθετε. Δηλαδή, επί της προτάσεως που από ό,τι κατάλαβα είπατε ότι αυτά τα πρωτόκολλα και οι στόχοι των πρωτοκόλων να μπορέσουν τελικά να επιτευχθούν μέσω άλλης οδού μέσω της κοινωνίας των πολιτών ίσως και βλέπουμε υπάρχει πλούτος σχεδίων βούλησης ε, προγραμμάτων διότι ανακαλύπτοντας τον άλλο ανακαλύπτει κανείς τον εαυτό του και οι Τούρκοι ανακαλύπτουν ε, τον ε, άλλον, την άλλη πλευρά του, την αρμενική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και προγράμματα που είναι επωφελή οικονομικά κιόλα. Άμεσα αποτελέσματα σε αυτά τις σχέσεις οικονομικές στον τομέα της συνεργασίας Αναφέρατε κάποια θέματα, την ασφάλεια, την υγεία, τον τουρισμό κλπ. Και επ' αυτής της βάσεως, της πολύ ρεαλιστικής, της πραγματιστικής, μπορούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που θα ευνοούσαν αυτές τη δημιουργία νέων σχέσεων. Ο καθένας υπογράμμισε, όλοι οι συνάδελφοι, ότι είναι σημαντικό, είναι κεφαλαιόδου σημασία για το μέλλον και για την περιφέρεια. Άρα, εδώ τίθεται το εξή θέμα οι τα περιφερειακά προβλήματα θα βαρύνουν και θα παγώσουν τη διαδικασία εξομάλυνσης για τη συμφιλίωση ή αντιθέτως συγκεκριμένες πρόοδοι όσον αφορά τα προβλήματα Τουρκίας-Αρμενίας μήπως η αντιμετώπιση τους ανοίγει προοπτικές θετικές για την ίδια την περιοχή όπως το θέμα το κουρδικό, το θέμα της Συρίας Προφανώς το θέμα της Ρωσίας είναι σημαντικό, πολλοί το ανέφεραν συνάδελφοι, αναφέρθηκαν στο ρόλο της Ρωσίας. Είναι αποφασιστική σημασία να εξεταστεί αυτό. Αυτά τα θέματα, επ' αυτών, τίθεται η περιφερειακή τραγωδία, θα έλεγα. Δεν είναι ώρα για συμπεράσματα, διότι όπως έλεγε κάποιος από τους προσκεκλημένους, δεν υπάρχουν συμπεράσματα που μπορούμε να συναγάγουμε σε αυτό το στάδιο. Ήδη θέλω να συγχαρώ. Ε, σας συγχαρώ για την εξαγωγή της συζήτησης, για το ενδιαφέρον σας. Και υπήρξαν και κάποιες πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν. Και ίσως η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πώς να το πω, δεν βρίσκω τις λέξεις μου. Μήπως είναι υπερβολικά αισιόδοξο να λέμε ότι θα μπορούσαμε να, να καλέσουμε εδώ συναδέλφους της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης, της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ξανασυζητήσουμε ε, τα θέματα που συζητήθηκαν εδώ. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και ίσως θα μπορούσε να μεταδοθεί και στο διαδίκτυο. Όπως και τώρα γίνεται, δεν τον έφερα στους παριστάμενους παρακολουθούν ε, οι ενδιαφερόμενοι τη συζήτηση μέσω διαδικτύου αυτή τη στιγμή. Ποια σειρά θέλετε να ακολουθήσετε. Εσείς ξεκινάτε. Ωραία, πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω ακολουθώντας το πνεύμα που επικρατεί σε αυτή την αίθουσα. Κάθε ερώτηση, ανεξάρτητα από αυτές με τις οποίες ε, διαφωνώ ε, κάθετα και με εκείνες με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα, είναι ειλικρινής και αξίζουν ειλικρινή απάντηση και στην πραγματική πιθανότητα να γίνω ε, ε, πολύ λίγο δημοφιλής στο Γερεβάν, τον Μπακού και στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω ειλικρινά σε κάθε ερώτηση. Λοιπόν, Αρμενία, Τουρκία, μετά Ναγκόρνο, Καραμπάχ. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ανέφερα τη Ρωσία επανειλημμένα, αλλά για να το θέσω καθαρά, η εξομάλυνση, προσπάθεια εξομάλυνσης αφορά Άγκυρα Γερεβάν. Όχι Άγκυρα Γερεβάν και την αρμενική κοινότητα του Glendale Καλιφόρνια ή τον Πακού. Πρόκειται περί διμερούς προσπαθίας εξομάλυνσης, όχι συμφιλίωσης. Είναι ένα πρώτο βήμα και για να είμαι ειλικρινής, αν δούμε την πολιτική των ΗΠΑ ή τη ρωσική πολιτική όσον αφορά αυτό το θέμα, και οι Αμερικανοί, ακόμα και οι Ρώσοι συμφωνούν ότι το μπαλάκι είναι ε, στο γήπεδο της Τουρκίας. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας το παιχνίδι ποδοσφαίρου. Το βάζουν περισσότερο στην Τουρκία από ότι στην Αρμενία. Πολλοί στην αρμενική κυβέρνηση εξακολουθούν να περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο από την Άγκυρα, να του πάρουν τηλέφωνο από την Άγκυρα. Όμω, όπω βλέπουμε εμεί τα πράγματα, υπάρχουν πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθεί ένα πολιτικό περιβάλλον που θα δικαιολογεί μια επιστροφή σε διπλωματικέ προσπάθειε. Γι' αυτό λοιπόν να στραφούμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όπω είπα δημοσία και σαφώς τον Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν είναι πλέον α, προεπετούμενο για την εξομάλυνση. Πράγματι αληθεύει. Όμως έμεσα βεβαίως τον Αγκόρνο Καραμπάχ αποτελεί ένα κομμάτι του πακέτου. Δεν θα προσβάλλω την ευφυΐα σας λέγοντας το αντίθετο. Αλλά αυτό που αντικατοπτρίζει είναι και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όπως την αξιολογώ εγώ. Αν η εξομάλυση σχέσεων ε, Αρμενίας-Τουρκίας ξεκινήσει τώρα, ξαναρχίσει τώρα και άγκυρα καλέσει τον πρέσβη και ξεκινάμε. Ακόμα και σε αυτή την καλύτερη περίπτωση, οποιαδήποτε πρόοδος για τον Αγκόρνο Καραμπάχ θα γίνει πιο δύσκολη και θα απομακρύνεται. Για την αρμενική κυβέρνηση συμβιβασμός και ένα άνοιγμα για τη σχέση με την Τουρκία θα ήταν κάτι πολύ μεγάλο για να μπορέσουν να στραφούν προς τον Αγκόρνο Καραμπάχ αμέσως. Μετά, το αντίθετο, χειρότερη περίπτωση. Δεν ξανανοίγουμε ποτέ τα σύνορα και δεν αποκαθίσταται διπλωματικές σχέσεις ποτέ. Και αυτό επιβεβαιώνει απλώς τη θέση και την εξουσία των σκληροπυρηνικών εθνικιστών και στις δύο χώρες μας, που θα μας θεωρήσουν ότι όλοι μας είμαστε αφελείς, καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση ότι είμαστε προδότες. Και γι' αυτό από μια ευρωπαϊκή έποψη των πραγμάτων το κλειδί είναι να δώσουμε την εξουσία, τη δύναμη στους μετριοπαθείς και όχι στους ακρεφνείς. Και πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχει στατιωτική λύση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πιο συγκεκριμένα, για να, είμαστε, για να είμαι ειλικρινής, με τον κύριο Νταβούτογλου και τον πρόεδρο Γκιούλ συναντήθηκα δύο φορές. Από τουρκική πλευρά θέλουν να είναι εξαιρετικά ευέλικτοι όσον αφορά τον ορισμό της προόδου από την πλευρά της Αρμενίας. Παραδείγματο χάρη, εγώ συνέστησα στην αρμενική πλευρά μονομερή απόσυρση ε, των ε, ελευθέρων σκοπευτών. Ε, θα ήταν μονομερής επίδειξη καλή θέληση και να αποκλιματοθεί η ένταση και να μειωθεί ο κίνδυνος πολέμου από κάποιο ατύχημα μέσω μικροσυγκρούσεων που ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Και τα καλά νέα είναι ότι η πολιτική ανεπίσημη και επίσημη της κυβέρνησης Αρμενίας θεωρεί τις υποκατοχήν περιοχές, περιοχές σαν υποκατοχήν. Στο Γέρεβαν υποκατοχήν, όχι απελευθερωμένος. Θα το θεωρούσαν αυτό ότι είναι σαν ένα χαρτί για διαπραγμάτευση και ότι πρέπει να επιστραφούν οι κατεχόμενες περιοχές. Είναι ζήτημα προς διαπραγμάτευση. Εκεί τίθεται σε ποιο βαθμό και σε ποια φάση οι κατεχόμενες περιοχές μπορεί να επιστραφούν. Πρέπει να δοθούν εγγύσεις για την ασφάλεια. Είναι βασική σημασία. Ναι. Ταυτόχρονα όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσον αφορά την πόλωση το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ομάδα του Μίνσκ παρόλο που θέλω να συμμετέχει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα του ε, Μίνσκ είναι απλώς διαμεσολαβητής. Μπορεί να κάνει αυτά που τα αντικρουόμενα μέρη μπορούν να κάνουν και θέλουν να κάνουν. Με άλλα λόγια, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η γενική έλλειψη πολιτικής βούλησης είναι ένα από τα τρία θεμελιώδη ε, ομπόδια για τη λύση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεύτερο εμπόδιο, αγνοούμε τα μαθήματα από τους Ιρλανδούς και, τις, ε, και των Βρετανών, Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Επί χρόνια οι Βρετανοί αρνήθηκαν και ανακαθέσουν να συνομιλήσουν με το συμφέινι το ΑΡΕΙ στα πλαίσια τη Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Και, και οι δεν συνομίλησαν με την οργάνωση στην απελευθέρωση τη ε, Παλαιστίνη. Μόνο όλα τα μέρη ήρθαν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, σαν συμμετέχοντε στην κρίση, μόνο τότε μπορούσε να επιτευχθεί η συμφωνία. Το Ναγκόρνο, Καραμπάχ δεν συμμετέχει άμεσα στην ειρευτική διαδικασία, στι διαπραγματεύσει. Και δεν θέλω να προσβάλλω την Αρμενία, αλλά ποιο έδωσε στην Αρμενία το μονοπόλιο των διαπραγματεύσεων εκ μέρου του. Και πιο σημαντικό, γιατί το Αζερμπαϊτζάν επιμένει και δεν διαπραγματεύεται άμεσα με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Ρίστο εν παρόδο έχει, είναι πιο δημοκρατικό, έχει πιο ελεύθερε εκλογέ από το Αζερμπαϊτζάν ή η Αρμενία. Τον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι πιο ελεύθερο. Ε, ταυτόχρονα είναι μια οδέτερη προσέγγιση που θα μπορούσε να ε, εφαρμοστεί. Ε, δεν δημιουργείται κάποια εξάρτηση αν ξεκινήσει ο διάλογος. Και μετά τρίτο, για να είμαστε ρεαλιστές, και οι δύο πλευρές, ή μάλλον και οι τρεις πλευρές αν θέλετε, βλέπουν αυτή την σύγκρουση από διαφορετικές οπτικές γωνίες για τα Τζερμπαϊτζάν. Θεωρούν ότι χάσαν την μάχη αλλά δεν έληξε ο πόλεμος. Για τους Αρμενίους είναι η πρώτη στρατηγική νίκη μετά από 2.000 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να επαναχωρήσουν μετά από αυτό. Και ο πόλεμος έληξε από την αρμενική πλευρά. Έτσι δε περαιτέρω, αν δούμε τη διπλωματική στρατηγική εγώ λέω ότι η διπλωματική στρατηγική του Αζερβαϊτζάν δεν είναι ούτε διπλωματική ούτε στρατηγική. Αυτή είναι η επίκρισή μου. Είναι μαξιμαλιστική. Θέλει τα πάντα και άλλα. Και για να είμαι ειλικρινή, βαρέθηκα να ακούω κατηγορίε ότι η Αρμενία κατέχει ε, την Αφροδίτη το φεγγάρι. Δεν είμαστε τόσο φιλόδοξοι να πάμε από ωκεανό σε ωκεανό και από θάλασσα σε θάλασσα. Η Αρμενία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που θέτει στετιωτική απειλή για κανένα. Δεν είναι στετιωτική απειλή για κανένα και η μόνη χώρα που συμβάλλει σε περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αλλά ποια είναι η επίκρισή μου. Γενικά η έλλειψη ηγεσία. Η Αρμενία με την απόφαση για τελωνιακή ένωση δημιουργεί τον κίνδυνο για την Αρμενία να απομονωθεί. Τα σύνορα θα ανοίξουν ποτέ ξανά και θα γίνει ασήμαντη. Αυτή είναι η απειλή. Κανεί δεν θα νοιάζεται πια για την Αρμενία ε, εκτός από τη διασπορά. Αυτή είναι η απειλή. Να γίνει ίσως μια χώρα στην πρώτη γραμμή ε, φρούριο της Ρωσίας. Παραπέρα, άμα δούμε τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ε, πρέπει η πρόοδος να γίνει για να δικαιολογηθεί η επιστροφή στη διπλωματία, όλες πλευρές να γίνουν πιο δημιουργικές και πιο ευέλικτες. Το πρόβλημα, και λυπάμαι την τουρκική πλευρά, είναι μεγάλη, ισχυρή, με μεγάλη οικονομική ισχύ. Έτσι έχει γίνει η Τουρκία, αλλά είναι ο όμοιρος του γιου πρώτερου ηγέτου του Αζερμπαϊτζάν που κληρονόμησε τη θέση λόγω γονιδίων και μπορεί να ευνοήσει και να στηρίξει και να καταστρέψει τις επιλογές διπλωματικές της Τουρκίας. Εγώ λυπάμαι την τουρκική πλευρά, για να είμαι ειλικρινής, στρεφόμενος προς την Ουάσιγκτον από αμερικανική έποψη. Δεν μιλώ εκ μέρους της αμερικανικής και με, μετακόμισα στην Αρμενία εδώ και 8 χρόνια ενώ ήταν ηγέτης τότε ο Cowboys ο Bush, είμαι δημοκράτης, μου αρέσει ο Ομπάμα αλλά δεν υπάρχει αμερικανική πολιτική στην περιοχή είναι υποσύνολο των σχέσεων Αμερικής-Ρωσίας, είναι υποπροϊόν της Τουρκίας και του Ιράν και πιο σημαντικό, εμείς ε, στη, από την ΙΠΑ φεύγουμε. Η ΙΠΑ αποσύρεται, μάλλον κλείνεται. Επιστρέφουμε. Είχαμε επεκταθεί υπερβολικά και σα, ρίχνουμε σε εσά το βάρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελπίζοντα ότι εσεί μπορείτε να καλύψετε το, το κενό τη απόσταση Αμερική και ίσω ε, ξεκινά και μια κάποια νέα σχέση και προσπάθεια να ξεκινήσει από την αρχή η σχέση μεταξύ Ρωσία ε, και ΗΠΑ. Λοιπόν, μην κοιτάτε προ εμά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην ευρύτερη περιφέρεια τη Ευρωπαϊκή Και στον Αγκόρνο Καραμπάκ, την τελευταία φορά που ε, ε, επεκτάθηκαν ήταν στο Key West το 2001 με το φίλο μου τον Κόλιν Πάουλ είχαμε πάει, ξέρετε τι έγινε, τι του συνέβη, αφού βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βασιστούμε στους Αμερικανούς. Η εξομάλυνση Αρμενίας-Τουρκίας των σχέσεων μπορεί να υποστηριχθεί από τους Αμερικανούς πώς, άμα εξαφανιστούν οι Αμερικανοί και να κάνουν οι άλλοι δουλειά τους. Εμείς δεν είμαστε εδώ να ικανοποιήσουμε τους Αμερικανούς, ούτε να φυσικάσουμε τους Ευρωπαίους. Μιλάμε για διμερή ιστορία. Δεν θέλω να προσβάλλω το Αζερβαϊτζάν, αλλά πραγματικά δεν ε, μπαίνεται εκτός του πλαισίου της γενοκτονίας και δεν θέλω να προσβάλλω τις άλλες χώρες, κυρίως τη Μόσχα. Α σταματήσω εδώ μου σταματάω εδώ. Okay. Quickly, five points. Σύντομα, πέντε ο θάνατος των πρωτοκόλων. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο έχουν παγώσει ως θανάτου, θυμούμενος θυμούμενο στην κρυογενετική που χρησιμοποιούν κάποιοι πλούσιοι Αμερικανοί για ε, να παγώσουν ε, το σώμα τους πριν ε, εκπνεύσουν τελείως και με την ελπίδα να μπορέσουν να επανέλθουν στη ζωή 50 χρόνια αργότερα. Ε, μένα μου θυμίζει αυτή η ιστορία του πρωτοκόλου το σχέδιο Ανάν, ξέρετε εάν ξαναγυρίσουμε την πρώτη γενιά συγκρούσεων της πρώτης τουρκικής κυβέρνησης, ακαπένου η ομιλητής, 2004-2007, και τις προσπάθειές της για την επίλυση των κρίσεων. Έχει τελειώσει όμως αυτό πια γιατί έχει ε, σε άλλες προσπάθειες, έχει καβαλήσει άλλα άλογα αυτή η κυβέρνηση. Και αυτά τα άλογα την πάνε αλλού, μακριά. Και αυτό άλλωστε το είπα και στην αρχή της ε, παρέμβασής μου, ότι έχει ε, αποδειχθεί σε μια προσπάθεια και ασχολείται αποκλειστικά με τη Συρία και λιγότερο με την Αίγυπτο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχει χρόνο και διάθεση για τίποτα άλλο. Επίσης, η δεύτερη οδός, ε, η οδός για το μέλλον και μου άρεσε η διατύπωση του Ρίτσαρτ που είπε ότι η δεύτερη οδός, το, το δεύτερο στάδιο ξεπερνάει την εξομάλυνση, γιατί η εξομάλυνση είναι ε, θέμα των, ε, πολιτών. Ε, το δεύτερο αυτό στάδιο σημαίνει συμφιλίου ουσιαστικά. Εκεί πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε, αλλά αυτό που δεν βλέπουμε ε, στην ιστορία όλη αυτή είναι ο παράγων Αζερβαϊτζάν. Και όσοι εδώ από το αξιόλογο κοινό που βρίσκονται γνωρίζουν κάπως καλύτερα την ε, κατάσταση θα διαπιστώνουν ασφαλώς ότι από την εικόνα αυτή λείπουν οι Αζέροι, οι ε, δημοκρατικές δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν. Άρα λοιπόν αυτό που οφείλουμε να πούμε και το, το σύστημα για τη σταθερότητα και νομίζω ότι θα φέρει αποτελέσματα γιατί και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ήδη έχουν ξεκινήσει τη δουλειά τους και με το είπα, θα έχουν, πιστεύω, με το μέσο σταθερότητα θα έχουν, πιστεύω, περισσότερε ευκαιρίε. Αλλά ελπίζω το προσεχέ είπα να συμπεριλάβει και την κοινωνία των Αζέρων. Για τα σύνορα. Ξέρετε, εμεί από το Ίδρυμα Χραντίνγκ έχουμε παραγγείλει μια οικονομετρική μελέτη για την εξέταση των συνεπειών του κλεισίματος ή του να μην το να ανοίξουν τα ε, σύνορα μεταξύ Τουρκίας και, Αρμένία. και Αρμενίας. Ομολογώ όμως ότι δεν μάθαμε τίποτα από τη μελέτη αυτή, γιατί το μόνο που έκανε ήταν να επαναλάβει δεδομένα και αποδείξεις προς, την, προς το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων. Οι περιοχές γύρω τα σύνορα αυτά οι παραμεθόριες περιοχές υποφέρουν πάρα πολύ από το ότι παραμένουν κλειστά. Το Κάρς είναι η πιο υπανάπτυκτη περιοχή της Τουρκίας και παραμένει. Επίσης, στα που είπε ο κύριος Βάικελ, για την ε, Τουρκία, για τη Ρωσία. Το έχουμε περιλάβει στην έκθεση και η ε, κυρία Φλότρου το ανέφερε επίσης. Ε, ο κύριος του παιχνιδιού εν προκειμένου στην περιοχή είναι η Ρωσία. Και προσπαθεί να διατηρήσει έναν έλεγχο μετά, τον ψυχρό, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Δεν μπόρεσε όμως η Τουρκία, παρά την αλλαγή των καταστάσεων, να εξασφαλίσει ισχυρό λόγο στην περιοχή. Ένα μονομε... Μια μονομερή κίνηση, το άνοιγμα των συνόρων από πλευρά Τουρκία. θα σήμαινε πιστεύω ένα ριζικό ε, βήμα που θα συγκλώνει τους Ρώσους και δεν θα καταλάβαιναν καν από πού τους ήρθαν. Και κάτι ακόμα σχετικό. Και ερώτηση περισσότερο προς όλους εσάς. Δινοηθείτε την Τουρκία ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης με προφανώς σύνορα ανοιχτά με την Αρμενία. Διανοηθείτε τι είδους συνέπειες που θα μπορούσε να φέρει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, ένα ελεύθερο εμπόριο στην περιοχή αυτή. Προφανώς πάρα πολλά θετικά και βέβαια αναλόγως θα κρυθεί και η μοίρα του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Αν συμφωνείτε μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας, να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας και όλους αυτούς που πήραν μέρος στη συζήτηση. Αν δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε, κυρίσω λοιπόν το τη συνεδρία Την επόμενη συνάντηση θα σας την ε, ανακοινώσει η Γραμματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και <laughs> τον τελευταίο λόγο θα το δώσω στην Ελένα. Ευχαριστώ πολύ Μίλαν. Λοιπόν, κλείνουμε τη συζήτηση αυτή που κατά την άποψή μου ήταν εξαιρετική βρήκαμε τους σωστούς εμπειρογνώμονες τα θέματα που θέσατε επιτάπητος ήταν ε, πολύ καλά βεβαίως σήμερα ήταν η πρεμιέρα ε, για τις συναντήσεις αυτής ε, αυτές θα προσπαθήσουμε και ο Μίλαν και εγώ να επαναλάβουμε τις συναντήσεις με το τέλος της θητείας μας για να βοηθήσουμε και εμείς αν είναι δυνατόν στη σύσφυξη των σχέσεων ε, Τουρκίας-Αρμενίας.